God Σας καλωσορίζω λοιπόν στην πρωινή μας συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε τις χθεσινές συζητήσεις. Σας καλωσορίζω όλους εγκάρδια. Έχουμε προσκαλέσει ορισμένους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα συζητήσουν τα θέματα τα οποία έχουμε από τις 9 μέχρι τις 11. Θα μιλήσουν για και θα σχολιάσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της γυναίκας και την καταπολέμηση του εγκλήματος των νέων. Η συγγήτρια ε, είναι η κυρία Άννα Ζαμπόρσκα η οποία θα παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας. Δυστυχώς έχει υπάρξει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα το οποίο σας έχει διανεμηθεί. Δυστυχώς ο δόκτωρ Κρίστιαν Φάιφα ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να είναι ο πρώτος ομιλητής, τον οποίο θα δίναμε το λόγο, δεν μπόρεσε να έρθει. Κολλείεται. Και έτσι δεν θα έχουμε την παρουσίαση του κυρίου Φάιφα. Πέραν τούτου, ελπίζω να μπορέσουμε να σεβαστούμε την ημερήσια διάταξη ως έχει. Και θα ξεκινήσω με την Άννα Ζαμπόσκα, την εισηγήτριά μας, που θα μας παρουσιάσει το κείμενο εργασίας της. Και μετά θα δώσω το λόγο, όπως είπα, στους εμπειρογνώμονες. Ελπίζω να γίνει μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, να σας καλωσορίσω και εγώ στην ακρόαση αυτή η οποία είναι αφιερωμένη στην εγκληματικότητα των νέων και στην συμβολή της πολιτικής ή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ισότητας ανδρών γυναικών και κατά πόσο συνεισφέρει στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας τους νέους. Ξεκινώντας θα ήθελα να θέσω ορισμένες ερωτήσεις. Αναρωτιέμαι, οι γονείς που είναι εδώ ξέρετε που είναι το παιδί σας αυτή τη στιγμή. Πού είναι. Οι πολιτικές ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της ε, ε, εγκληματικότητας στις μεγάλες πόλεις και πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της γονικής ευθύνης. Η Επιτροπή μας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής εντολής ασχολήθηκε με το θέμα και το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση της κυρίας Μπατζελή για την επιρροή, επιρροή συγγνώμη, την κοινωνική της γυναίκας στα κοινωνικά δρόμενα. Ο καθηγητής Φάιφα ήταν παρόν σε εκείνη την ε, ακρόαση την οποία είχαμε οργανώσει με αφορμή την έκθεση της κυρίας Μπατζελή και λυπάμαι που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η βία στους νέους είναι ένα φαινόμενο απειλητικό νέα παιδιά ασκούν βία και υπάρχει γενικά, μια, παρατηρείται μια αύξηση αυτής της μορφής της εγκληματικότητας. Η εγκληματικότητα αυτή και η βία είναι βασικό χαρακτηριστικό. Οι ξυλοδαρμοί, εκβιασμοί, βιασμοί και γενικά πολλές μορφές ε, ε, βίας. Ποιος είναι άραγε υπεύθυνο για την κατάσταση αυτή. Φταίνε οι εκπομπές της τηλεόρασης. Φταίει το διαδίκτυο. Φταίνε οι γονείς. Φταίει το σχολείο. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι, δείχνουν οι μελέτες, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι τομείς συγχωνεύονται θα έλεγα σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγον είναι η επιρροή του περιβάλλοντος όπως λέγαμε, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Και το δεύτερο ε, σημαντικός παράγοντας είναι ο χαρακτήρας του κάθε νέου. Για την προώθηση κάποιων πολιτικών υπάρχει μια χρόνια έλλειψη πόρων και πολλές φορές υπάρχει επίσης και μια δικαιολόγητη χρήση φυσικής τιμωρίας, σωματικής συγγνώμη τιμωρίας. Το έγγραφο αυτό βασίζεται, μάλλον το θέμα αυτό ε, είναι κάτι το οποίο προέρχεται θα έλεγα από την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη συμπεριφορά του νέου που πάρα πολύ συχνά αψηφά τους κοινωνικούς κανόνες και τις ε, πραγματικές υλικέ ε, συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν οι νέοι σήμερα και που επηρεάζουν την ανάληψη ευθυνών. Οι διάφοροι διεθνείς θεσμοί όπως ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζουν την βασική ευθύνη την οποία έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους και τα καθήκοντα των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Από την άλλη, η συμμετοχή των γονιών στην καταπολέμηση της παιδικής ή της νεανικής εγκληματικότητας είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ συχνά πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και στις συνθήκες, στις υλικές στα πλαίσια των οποίων μεγαλώνει το παιδί και πώς οι γονείς ασκούν τις αρμοδιότητές τους και, τις αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για να μην περάσω μετά στις διακρίσεις τις οποίες υφίστανται τα παιδιά όταν ξεκινούν να εργάζονται στο χώρο της εργασίας δεν θέλω να κατηγορήσω τους γονείς περισσότερο από όσο πρέπει, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι στο έγγραφό μου δεν έχω την πρόθεση να κατηγορήσω τους γονείς και να αποδώσω την κατάσταση αυτή μόνο στους γονείς. δεν πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι μόνο οι γονείς. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του παιδιού. Αυτό υπογραμμίζεται και στην έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας που προτείνει, κάνει μάλλον κάποιες προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των παιδιών σε μια πρώτη φάση σε πολλούς τομείς όπως τον οικογενειακό τομέα, τον κοινωνικό τομέα, τον σχολικό τομέα και γενικότερα τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης επιδεικνύοντας την απαιτούμενη αλληλεγγύη ανάμεσα στις διάφορες γενναίες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση και από των νέων, εμένοντας στην ευθύνη των γονέων, και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις βασικές συνθήκες ε, με τις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν πολιτικές εδώ λοιπόν, υπάρχουν είναι ερώτημα κάποιες πολιτικές ε, στις σχέσεις, που αφορούν τις σχέσεις ανδρών και γυναικών και που βοηθούν την καταπολέμηση της παιδικής εγκληματικότητας βοηθώντας τους γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Με άλλα λόγια, τι συνθήκες απαιτούνται έτσι ώστε να αποφύγουμε διακρίσεις και στον τομέα της αγοράς εργασίας και στις σχέσεις ανδρών γυναικών έτσι ώστε να παίζουν τον ρόλο τον οποίο έχουν στην ανατροφή των νέων παιδιών με σωστό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίες χαρακτηρίζουν θα έλεγα τις κοινωνικές συνθήκες που οδηγούν στην εγκληματικότητα των νέων και στη βία. Υπάρχουν τα φαινόμενα της αποσταθεροποίησης και της συναισθηματικής ακόμα αστάθειας στο εσωτερικό των οικογενειών. Θυμίζω ότι τα πρώτα θύματα της βίας που ασκούν οι νέοι είναι πολλές φορές εκτός από τους συνομιλίκους τους οι ίδιοι τους οι γονείς. Υπάρχουν επίσης και μακροοικονομικοί παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο λόγω ακριβώς της έλλειψης κοινωνικών μέτρων που οφείλονται σε δημογραφικά φαινόμενα Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη δημογραφία όταν εμείς προσπαθούμε να κατανοήσουμε την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα. Πολύ συχνά οι νέοι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, έχουν χάσει την πίστη τους στο μέλλον, έχουν χάσει την πίστη τους στο μέλλον της χώρας τους και αυτό τους αποσταθεροποιεί και αυτό προσπαθούμε να δούμε πώς τα διεθνή όργανα ε, αντιμετωπίζουν την σχέση ανάμεσα στην νεανική εγκληματικότητα και τις γονεϊκές ευθύνες. Η οικογένεια είναι πάντα η καλύτερη εγγύηση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στους νέους. Οι διεθνείς οργανισμοί προσπαθούν να συνδέσουν με κάποιο τρόπο τις γονεϊκές ευθύνες με την ανάπτυξη της εγκληματικότητας. Οι μελέτες από το 2003 στην Ευρώπη δείχνουν ποια είναι η κατάσταση σε επίπεδο εγκληματικότητας των νέων. Οι μελέτες του ΟΗΕ έχουν υπογραμμίσει τις τεράστιες ε, ευθύνες και τον τεράστιο ρόλο τον οποίο παίζει η οικογένεια. Από τις μελέτες του ΟΗΕ βλέπουμε ότι όταν υπάρχει αρκετή γονεϊκή ε, φροντίδα υπάρχει χαμηλή εγκληματικότητα. Οι δυσλειτουργικές οικογένειες που πολλές φορές συνδέονται με την έλλειψη γονεϊκού ελέγχου οδηγεί στην εγκληματικότητα πολύ συχνά όπως επίσης και η πρώιμη ανεξαρτητοποίηση των νέων και αυτή οδηγεί σε νεανική εγκληματικότητα. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει επίσης την σημασία που έχει η οικογένεια σε σχέση με τη βία και την υγεία. Οι γονεί, λέει ο Διεθνή Οργανισμό Υγείας, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη βίαιων συμπεριφορών στους νέους. Ιδιαίτερα στην εφηβεία. Η εμφάνιση φαινομένων βίας στην εφηβεία είναι κάτι το οποίο εν πολύ οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσαν τα παιδιά αυτά στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη έκθεσή του ε, έχει την λογική ότι η έλλειψη ε, κατανόησης ε, ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, η δυσλειτουργία των οικογενειών και πολλές φορές η απουσία των γονιών οδηγούν σε αύξηση των φαινομένων εγκληματικότητας στους νέους. Το θέμα της συζήτησης δεν είναι να αποδώσουμε απλά ευθύνες και να αρχίσουμε να κατηγορούμε τους γονείς. Αυτό που έχει σημασία είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων γενεών που θα πρέπει, των μελλοντικών γενεών συγγνώμη, που θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα σταματήσω εδώ με αυτές τις λίγες γενικές παρατηρήσεις, να ακούσω τους ακροατές και να μου επιτρέψετε να επανέλθω μετά. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζάμπορσκα για την εισαγωγική σας αυτή δήλωση. Μας μιλήσατε για το έγγραφο εργασίας που έχουμε. Τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας, τους εμπειρογνώμονες που βρίσκονται σήμερα εδώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένος. Εξού και ο καθένας από τους εμπειρογνώμονες έχει στη διάθεσή του 15 λεπτά. Θα ήθελα να δώσω καταρχάς το λόγο στην κυρία Γκούτρουν Νόρντμπορκ, η οποία είναι εμπειρογνώμων για θέματα φύλου στην Υπηρεσία Υποστήριξη Θυμάτων Εγκληματικών Ενεργειών στη Σουηδία. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή μας και περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε. Εκτός μικροφώνου. Uh, Θα ήθελα να πω ότι είναι περίπλοκα τα θέματα. Μάλλον να ξαναρχίσω, είχα κλειστό το μικρόφωνο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και που με ευθύνετε και την πρόσκληση. Λέγομαι Γκούντρουν Νόρντμπορκ, είμαι καθηγήτρια δικαίου. Βέβαια τώρα Εργάζομαι στην, ε, στον, στον ε, Σουηδικό Οργανισμό για την Υποστήριξη των Θυμάτων Εγκληματολογικών Ενεργειών. Από τη δεκαετία του 70 εργάζομαι στον τομέα των, σε, θέματα που έχουν να κάνουν με τους νέους. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ζαμπόρσκα για την ε, φιλοδοξία της σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νεανικής εγκληματικότητας. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και περίπλοκο, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σε όσο δυνατόν περισσότερα επίπεδα, σε παγκόσμιο, σε κοινοτικό και σε επίπεδο κρατών μελών. Βέβαια, η έρευνα την οποία εγώ γνωρίζω παρουσιάζει άλλες απόψεις ε, βασιζόμενοι σε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά τα οποία ακούσαμε από την κυρία Ζάμπροσκα θα πρέπει να δούμε ανάλογα με το που εστιάζουμε, δηλαδή στην ισότητα των φίλων ή στην οικογένεια, στη σταθερότητα της οικογένειας. Αν είναι σημαντικό να δούμε την ενδοοικογενειακή βία, για παράδειγμα, ή την ε, βία εκτός οικογένειας. Εγώ θα έλεγα και στις δύο περιπτώσεις. Θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα από την προσωπική μου εμπειρία για καλές πρακτικές και μεταρρυθμίσεις. Και θα ε, μιλήσω επίσης και για κάποιους γενικούς κανόνες, βασικούς κανόνες για όλους. Ποιο είναι το πρώτο ερώτημα, αν η ισότητα των δύο φίλων είναι σημαντικότερη από την οικογένεια. Δεν είμαι κατά της οικογένειας, φυσικά και όχι. Αλλά επειδή η ισότητα των δύο φίλων στην οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδίως για τα παιδιά, και είναι και σημαντική και για την ασφάλειά τους για να, έχουμε, για να υπάρχει σεβασμός προς αυτά αλλά και από αυτά προς τους άλλους. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επικεντρωνόμαστε σε μια ασφαλή και σταθερή οικογένεια ή σε μια σταθερή ή σε μια ασφαλή. Εγώ νομίζω ότι η σταθερή οικογένεια δεν είναι τόσο σημαντική όσο η ασφαλής οικογένεια. Επίσης, αν υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φίλων, μεταξύ των δύο συντρόφων, εντός εκτός γάμου, αυτό δημιουργεί πιο σταθερές οικογένειες. Αν λοιπόν τονίσουμε την ισότητα των δύο φίλων, θα έχουμε λιγότερους χωρισμούς, λιγότερα διαζύγια. Και βέβαια δεν θα υπάρχει βία αν υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φίλων. Αν δούμε τώρα την ενδοοικογενειακή βία. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη από αυτήν του εγγράφου εργασίας η οποία επικεντρώνεται στη βία εκτός της οικογένειας. Η οποία βία αυτή επηρεάζει την οικογένεια. Φυσικά και αυτό αληθεύει. Θα πρέπει όμως να δούμε την άλλη πλευρά, δηλαδή τη βία εντός της οικογένειας. Είμαι πεπισμένη ότι με την αστίαση αυτή μπορούμε να κάνουμε άλλες προτάσεις, διότι ανοίγονται νέες ε, προοπτικές. Η ανδρική βία είναι αυτή η οποία κυριαρχεί και εντός και εκτός της οικογένειας. Κυρίως ε, οι άντρε είναι αυτοί οι οποίοι ασκούν βία είτε στην σύζυγό του, συντροφό τους, είτε στα παιδιά τους μέσα στην οικογένεια. Και αυτή η βία έχει πάρα πολύ επιζήμια, πολύ επιβλαβή αποτελέσματα και στα παιδιά τα οποία γίνονται μάρτυρες αυτών των πράξεων βίας, ε, τα οποία ουσιαστικά εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν περιορίζεται αυτή η πράξη βίας μεταξύ των δύο συντρόφων. Πάντοτε σχεδόν τα παιδιά αντιλαμβάνονται, βλέπουν, γίνονται μάρτυρες ε, είτε ε, αυτόπτες είτε αυτοίκοοι αυτής της βίας. Και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που και το παιδί είναι το θύμα της βία, το πρωταρχικό. Αλλά τα αποτελέσματα είναι πάντοτε πάρα πολύ βλαβερά για τα παιδιά. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια βία οικογένεια οδηγεί επίσης και τα αγόρια να μάθουν και αυτά να χρησιμοποιούν τη βία ως ένα τρόπο ελέγχου. Και οδηγούν δηλαδή σε κάποιες πράξεις ε, που βίας για να εξασφαλίσουν την υποταγή των ε, τα κορίτσια μάλλον οδηγούνται στην υποταγή. Επίσης δημιουργείται μεγάλο ζήτημα και κοινωνικό και σε ό,τι αφορά την υγεία και βέβαια προκύπτει και σημαντικό κόστος για τους αμονωμένους, αμονωμένα άτομα και τις ε, κοινωνίες. Ό,τι αφορά τώρα τους ε, χωρισμούς και τα διαζύγια, θα πρέπει να τα υποστηρίζουμε και αν ε, ο βίαιος σύζυγος, ο βίαιος άντρας δεν συμφωνεί να ξεκινήσει κάποια θεραπεία για να αντιμετωπίσει την ανάγκη που έχει για κυριαρχία και άσκηση ισχύω. Επίση θα πρέπει να ενδυναμώσουμε και να υποστηρίξουμε τη θέση της μητέρα ω γονιού μετά από ένα διαζύγιο ή ένα χωρισμό γιατί τότε ενδέχεται πάλι να κινδυνεύουν τα παιδιά. Και αν μετά από μια σχέση βίαιη ε, που έχει οδηγήσει σε χωρισμό θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι θα χρειαστεί και οικονομική υποστήριξη και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πάρα πολύ κακές εμπειρίες ε, που είχαν από, λόγω της βίας η μητέρα και τα παιδιά. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι επίκεντρο της προσοχής. Και βλέπουμε και από την έρευνα ότι οι μονογονικές οικογένειες επίσης ε, κάποιες φορές ε, υπάρχει ένας κίνδυνος και για το παιδί. Ποιον θα πρέπει να κατηγορήσουμε γι' αυτόν, ε, τη, τη μητέρα που την τη μόνη στην οικογένεια ή τον βίαιο άντρα. Και θα πρέπει να βλέπουμε και να υποστηρίζουμε τη μη βία πλευρά της οικογένειας. Θα μιλήσω τώρα για κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις και καλές πρακτικές. Πρώτα απ' όλα, αποκλεισμός, απαγόρευση μάλλον, Τη σωματική τιμωρία ή αν όχι ακριβώ απαγόρευση, τουλάχιστον αντιμετώπιση καταλέμη τη μέσα στην οικογένεια. Εγώ θα πρώτε να βέβαια ή αν όχι ακριβώς απαγόρευση, τουλάχιστον ε, αντιμετώπιση, καταπολέμησή τη μέσα στην οικογένεια. Εγώ θα πρότεινα βέβαια απαγόρευση τη σωματικη ε, τιμωρια Το 1979 η Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα που το έκανε. Τώρα περίπου 25 χώρες έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα της Σουηδίας. Και ο ΙΕ υποστηρίζει και ενθαρρύνει και άλλους να συμμετάσχουν. Και από την παγκόσμια έρευνα ε, βλέπουμε ότι είναι η σημαντικότερη δράση για την πρόληψη της εγκληματικότητας, η απαγόρευση σωματικής τιμωρίας. Εξίσου σημαντικό βέβαια είναι να συζητήσουμε και να επικεντρωθούμε σε κάποιες εναλλακτικές μορφές, σε κάποιους εναλλακτικούς τρόπους για την επίλυση των ε, συγκρούσεων. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι η γονική άδεια είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση και καλό θα ήταν να υπάρχει εξίσωση ε, χρονική σε ό,τι αφορά και τη μητέρα και τον πατέρα. Νομίζω ότι η μητρότητα είναι μια υποχρέωση. Υπάρχουν σημαντικοί κανόνες που ισχύουν για τη μητέρα, αλλά η πατρότητα φαίνεται να είναι κάπως ε, πιο προερωτική αν θέλετε ή εθελοντική. Αλλά νομίζω ότι και τους πατεράδες πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να είναι καλοί στο ρόλο τους, στο ρόλο του γονιού. Θα συνεχίσω με τα ζητήματα του φίλου, αλλά σε άλλα επίπεδα τώρα. Παιδική μέρημνα, σχολεία, πανεπιστήμια. Πρέπει να δούμε δηλαδή πάρα πολλούς τομείς. εάν υπάρχουν κάποιοι νέοι οι οποίοι διαπράττουν ε, εγκληματικέ ενέργειε, εγώ νομίζω ότι μια δυνατότητα είναι η διατησία, η διαμεσολάβηση. ώστε να μάθει, να καταλάβει ο νεαρός παραβάτης ε, τι επιπτώσεις είχαν οι πράξεις του ή έχουν οι πράξεις τους οι νεαροί παραβάτε πρέπει να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίε. Αυτού κυρίω επικεντρωνόμαστε εμεί. Και αν αυτό ο νεαρό παραβάτη διαπράξει μια αξιόπινη πράξη και είναι πρόθυμο να στήσει γνώμη στο θύμα και μετά να ακούσει και να κατανοήσει τα αποτελέσματα της ε, πράξης του, θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Και βοηθά στην καταπολέμηση της ε, εγκληματικότητας. Θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω μία πρόταση του επικεφαλής της υπαρχιακής αστυνομίας της Στοκχόλμης που λέγεται Project Boy για την αποφυγή εγκληματικών ενεργειών από αγόρια. Είναι η πρώτη φορά που τίθεται ως πρόβλημα η αρενοπότητα, αν θέλετε, ως στερεότυπο και αναλαμβάνονται σχετικές δράσεις. Η αρενοπότητα, η υπερβολική επίδειξη του ανδρισμού είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια κάποιες φορές που άνδρας είναι ο κανόνας, εκεί δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό ως πρόβλημα. Κυριαρχούν σε όλες τις αστικές οι άνδρες και, και τα αγόρια και στην νεανική εγκληματικότητα. Τα νεαρά αγόρια είναι αυτά που στο πολύ μεγάλο ποσοστό τους, ε, όχι τα νεαρά κορίτσια, κάνουν τις εγκληματικές αυτές ενέργειες μεταξύ των νεαρών παραβατών. Εάν συνδυάσουμε Πάντως αν δούμε γενικώ την κατάσταση δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Μια εναλλακτική λύση ενδεχομένω θα ήταν ε, ένα γυναικείο πρότυπο κατά κάποιο τρόπο. Ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να ενδυναμωθεί είναι το πλαίσιο της ε, ζωής της γυναίκας που θα πρέπει να έχει νομικά δικαιώματα. Είτε αυτά ασκούνται από άνδρες είτε από γυναίκες και με αυτή τη βάση αυτό το γυναικείο πρότυπο είναι αυτό που πρέπει να θεσπιστεί και να ενισχυθεί από κοινού και σε ίδιο επίπεδο με το πλαίσιο της ζωής του άντρα. Αυτό έχει πει ένας ερευνητής. Μια άλλη, ο Τόφ Σταγκντάλ και μια άλλη ερευνήτρια από τις ΗΠΑ, η Κάθρε Μακίνον, λέει ότι πριν από κάθε, μάλλον πίσω από κάθε νόμο μπορούμε να βρούμε τις ε, εμπειρίες ζωής κάποιου διότι ποτέ δεν προηγείται ο νόμος της ζωής. Πάντα προηγείται η ζωή. Το θέμα λοιπόν ε, και το ερώτημα και στην πολιτική και στην ιστορία αλλά και στο δίκαιο και στο νόμο είναι ποιου οι εμπειρίες δημιούργησαν δύσκολους ε, διαφορετικούς ε, νόμους. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε μεταξύ άλλων, όπως σας είπα, στις εμπειρίες των γυναικών, περισσότερο από ό,τι το κάνουμε μέχρι τώρα και επίσης να ακούσουμε πιο προσεκτικά και τις εμπειρίες των παιδιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Νόρτμπορκ για την ε, συμβολή αυτή στη συζήτηση. Ευχαριστούμε και πάλι και προχωρούμε στο πρόγραμμα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ελίζα Μάνα, διευθύντρια του τμήματος ε, πολιτιστικής πολιτικής στην Ιταλία, του Σένσης, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Σβένσον. Φροντίζω τον τομέα έρευνας του Τσένσης, οργάνωση που ασχολείται με νέους, γυναίκες, μέσα ενημέρωσης και πολιτιστικές πολιτικές γενικότερα. Άκουσα κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις για την επιρροή που παίζουν κάποιες υπηρεσίες κοινωνικοποίησης τους νέους. Σχετικά με τη δική μου χώρα, έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το σύστημα των μέσων ενημέρωσης και το περιεχόμενο λεγόμενων ΜΜΕ εδώ και 30 περίπου χρόνια επηρεάζει ιδιαίτερα θα έλεγα την εικόνα της γυναίκας στην Ιταλική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 οι γυναίκες στην Ιταλία είχαν πετύχει πάρα πολύ σημαντικά θετικά βήματα αλλά η σημερινή τηλεόραση στην ουσία κυκλοφορεί μια εικόνα της γυναίκας ιδιαίτερα στερεοτυπική. Εμείς στην οργάνωση Τσένσης και μετά από τη συνεισφορά της κυρίας Κώστα έχουμε κυκλοφορήσει μια λευκή βίβλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ονομάζεται «Γυναίκα και Μέσα Ενημέρωση στην Ευρώπη». Το έγγραφο αυτό δείχνει πως αντίθετα με αυτά που συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν κώδικες αυτορύθμισης, νόμοι και ορθές πρακτικές για την προώθηση στην τηλεόραση και στα μέσα ενημέρωσης μια εικόνα των γυναικών που να είναι πραγματική, που να είναι αντίστοιχη με την καθημερινότητα των γυναικών, που να δείχνει τις γυναίκες για αυτό που είναι πράγματι, έτσι όπως ε, έχουν αναπτυχθεί στις σπουδές ε, στον επαγγελματικό χώρο και στη συνεισφορά τους στον κοινωνικό τομέα. Δυστυχώς όμως αυτό στην Ιταλία και στην Ιταλική τηλεόραση δεν συμβαίνει. Η εικόνα της γυναίκας συνδέεται ε, με κάποια στερεότυπα σεξουαλικά. Ονομάζουμε αυτό το πράγμα στην Ιταλία το φαινόμενο της γλάστρας, όπως λέμε στην Ελλάδα. Πάρα πολλές γυναίκες, ημίγυμνες, οι οποίες δεν ομιλούν ποτέ και που στολίζουν, θα έλεγα, όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα σε όλες τις ώρες της ημέρας. Αυτό επηρεάζει φυσικά τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλλα, ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Τώρα σας τα λέω αυτά κάπως υπεραπλουστευτικά για λόγους χρόνου. Οι παράγοντες είναι πολλοί, το διακύβευμα είναι μεγάλο, αλλά είναι προφανές ότι μία συνεχής ενημέρωση που παρουσιάζει τη γυναίκα συστηματικά σαν σεξουαλικό αντικείμενο δεν μπορεί παρά να στρεβλώνει τις σχέσεις της διαγενεϊκές. Στα πλαίσια των σχέσεων αυτών η αξιοπρέπεια της γυναίκας σαν πρόσωπο συστηματικά σκιάζεται και αγνοείται. Και αυτό φυσικά επηρεάζει και στο εσωτερικό, τη σχέση στο εσωτερικό των οικογενειών, τη σχέση σε εισαγωγικά εξουσίας ανάμεσα σε, στους δύο συντρόφους, ανάμεσα στους δύο συζύγους. Επηρεάζει επίσης και τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια στο εσωτερικό της ίδιας οικογένειας, αλλά και εκτός οικογένειας, σε κοινωνικούς χώρους. Η εικόνα την οποία δείχνουν για τις γυναίκες η ελίτ της χώρας είναι πάρα πολύ εύκολο μια γυναίκα να μπορέσει να πετύχει το όνειρό της να ασκήσει ένα κάποιο επάγγελμα βέβαια. Οι γυναίκες γιατροί στην Ιταλία είναι περισσότερες από τους άνδρες ιατρούς. Έχουμε πετύχει πολλά. Αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο οι γυναίκες να κάνουν μια στραδιοδρομία υψηλού επίπεδου, να αποκτήσουν θέσεις ευθύνης, Ακριβώς γιατί η εικόνα της γυναίκας είναι μια εικόνα δευτερεύουσα, συμπληρωματική της αντίστοιχης του άνδρα. Με ποιο τρόπο λοιπόν η κατάσταση αυτή μπορεί να συνεισφέρει στα φαινόμενα βίας. Πάρα πολύ απλό είναι. Όρια έχουν συνηθίσει να θεωρούν τις γυναίκες σαν σεξουαλικό και μόνον αντικείμενο και όχι σαν ένα πραγματικό πρόσωπο. Αυτό δημιουργεί στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στις συντρόφους και στις γυναίκες, στις συνομήλικες ή όχι γενικότερα. Υπάρχουν φαινόμενα α, βίας εις βάρος ενήλικων γυναικών από πλευράς ανηλίκων. Λοιπόν, έχουν ε, μια αντίληψη για τη γυναίκα χρηστική και όχι πραγματικής σχέσης ανάμεσα σε δύο πρόσωπα ισότιμα. Αυτό μας ανησυχεί λοιπόν, μας ανησυχεί πολύ. Οι προσεκτικοί παρατηρητές στην Ιταλία ανησυχούν γιατί πρόκειται για μια διαδικασία η οποία κρατά εδώ και πάρα πολλές ε, δεκαετίες. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει θα έλεγα διαπεράσει και χαρακτηρίσει την συλλογική νοοτροπία. Εγώ είμαι μέλος μιας κυβερνητικής επιτροπής, η οποία ονομάζεται Μέσα Ενημέρωσης και Ανήλικη και θα έπρεπε να προστατεύει τους νέους, τους ανηλίκους από τις αρνητικές επιπτώσεις της τηλεόρασης. Έχουμε τεράστιες δυσκολίες, παρά όλη την καλή θέληση την οποία επιδεικνύουμε, έχουμε τεράστιες δυσκολίες για να λειτουργήσουμε, γιατί θα πρέπει να λογοκρίνουμε ουσιαστικά το 70% των προγραμμάτων τα οποία εκπέμπονται. Συνεπώς λοιπόν μας δημιουργείται η αίσθηση ότι είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι σε σχέση με το τεράστιο μέγεθος που έχει αποκτήσει το πρόβλημα. Ως εκ τούτου λοιπόν η αναφορά για μας είναι κάτι το θεμελιώδες. Η Λευκή Βίβλος στην οποία αναφέρθηκα έχει κυκλοφορήσει πολύ και στο εξωτερικό έχει εξαντληθεί το έγγραφο αυτό και είχε εγγραφτεί ήδη το 2005 και θα ήθελα να το επικαιροποιήσω ακόμα για να δείξουμε στην Ιταλία πόσο εμείς έχουμε μείνει πίσω. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε έναν πολιτισμό για την εικόνα των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης γιατί κάτι τέτοιο επηρεάζει άμεσα τις συμπεριφορές των νέων ανθρώπων. Θα ήθελα επίσης να σταθώ σε ένα ειδικό θέμα που είναι οι διαφημίσεις που βλέπει κανείς στο δρόμο. Εγώ γυρνώ στην Ευρώπη, ταξιδεύω σε πολλές χώρες και δεν έχω δει πουθενά αλλού εκτός από την Ιταλία μια τόσο στρεβλή και παραποιημένη εικόνα της πραγματικότητας όσο στην Ιταλία. Αυτό γιατί δυστυχώς οι γενικές επιθυμίες πηγαίνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό το οποίο που σε μία άλλη χώρα θα σας έκανε να σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής σας, στην Ιταλία θεωρείται κάτι το πάρα πολύ φυσικό και συνηθισμένο. Αυτό είναι λοιπόν το φαινόμενο το οποίο ορισμένοι παρατηρητής, μεταξύ των οποίων και εγώ ιδία, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε. Και σε συνεργασία με τη Σίλβια Κώστα έχουμε απευθύνει και μια έκκληση στον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να παρέμβει και να μας βοηθήσει να προωθήσουμε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις και αναφέρομαι εδώ στον νόμο ο οποίος καθορίζει τη σχέση ανάμεσα στη δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο. Να προφήσει λοιπόν κάποιες νομικές ρυθμίσεις που να περιλαμβάνει κάποιες τροπολογίες υπέρ της προστασίας της αξιοπρέπειας της γυναίκας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία αναφορά που αναφέρεται στην αξιοπρέπεια της γυναικείας εικόνας. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι το θέμα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας και τη χώρα μας. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας κάνει να αλλάξουμε πορεία. Η βία εις βάρος των γυναικών δεν είναι μόνο η βία η προφανής. Εγώ έχω ε, στοιχεία σχετικά με τις εγκληματικές πράξεις ε, που διαπράττονται από τους νέους. Αλλά η βία δεν είναι μόνο αυτή. Μιλάμε επίσης και για την ελαφρία άσκηση βίας που συμβαίνει σε καθημερινή βάση. Η συνάδελφος έλεγε ότι πρώτα συμβαίνει το φαινόμενο το φυσικό, πρώτα έρχεται η ζωή και μετά ο νόμος. Και ο νόμος είναι συνέπεια ουσιαστικά των συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν την πραγματική ζωή. Είναι λοιπόν απαραίτητο να προσπαθήσουμε έστω και σε μία πρώτη φάση ερευνητικά να εντοπίσουμε αυτές τις ε, πράξεις της λεγόμενης μικροβίας. Γιατί η βία δεν είναι μόνο η, βία η έντονη πράξη που προκαλεί σωματική βλάβη, αλλά υπάρχει καθημερινή άσκηση βίας, λεκτική βία. Σε μια γυναίκα λέει κανείς κάτι το οποίο δεν θα έλεγε σε έναν άνδρα στην ουσία σε μια γυναίκα ε, της αφαιρεί κανείς πάρα πολύ εύκολα το λόγο από ότι σε ένα αγόρι ή σε έναν άνδρα. Συνεπώς λοιπόν υπάρχουν στερεότυπα θα έλεγα τα οποία είναι υποβόσκοντα, αποκεκριμένα, τα οποία θα πρέπει να έλθουν πλέον στην επιφάνεια. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, έτσι ώστε να δείξουμε τα ποιοτικά, ψυχολογικά χαρακτηριστικά, για να μην πω και ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά του θέματος. Γιατί πίσω από μια βίαιη συμπεριφορά υπάρχει πάντα και μια αντίληψη για τη βία, που συνδέεται στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα στερεότυπα που επιβάλλουν οι άνδρες. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ελπίζω να συνεχιστεί η ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάνα για την παρέμβασή σας στη συζήτησή μας σήμερα και δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Μάρκο Περολίνη ο οποίος είναι υπεύθυνο πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας στο Βέλγιο. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και την κυρία Ζαμπόρσκα για το έγγραφο εργασίας και την παρουσίασή της. Τρία-τέσσερα σημεία θέλω να αναπτύξω στην ομιλία μου Πρώτον, θέλω να εξηγήσω ποια είναι η αιτιακή σχέση μεταξύ μεμονωμένων παραγόντων, οικογένεια, γονική ευθύνη και ε, νεανική εγκληματικότητα και πώς υπερεκτιμάται, ενώ οι κοινωνικοί παράγοντες υποτιμώνται. Μετά θα μιλήσω για τη σχέση μεταξύ φύλου και εγκλημάτων αδικημάτων των νέων και τέλος κάποιες ε, πολιτικές δράσεις και λύσεις που μπορούμε να προτείνουμε. Σύμφωνα με την άποψή μας στο έγγραφο εργασίας δεν, επηρεάζει, δεν, δεν λαμβάνει υπόψη κοινωνικούς παράγοντες όπως διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό, ούτε λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα ε, αδικήματα δεν είναι προβλέψιμα και η νεανική εγκληματικότητα δεν είναι πάντα προβλέψιμη και δεν συνδέεται πάντα με παράγοντες κινδύνου Υπάρχουν πολλές έρευνες που επικεντρώνουν στην ε, σχέση και σύνδεση μεταξύ γονική ευθύνη και έγκλημα, αλλά από την άλλη υπάρχουν και πολλές έρευνες που αμφισβητούν την αιτιακή σχέση μεταξύ των δύο αυτών. Για παράδειγμα, ε, ο Οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεμελιώδη δικαιώματα, έκανε μια έρευνα μεταξύ αυτών που είναι νέοι που υφίστανται διακρίσεις, κοινωνικό, κοινωνική περιθωριοποίηση και βία και σύμφωνα με αυτή τη μελέτη υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ διακρίσεων κοινωνικού αποκλεισμού και βίας. Εκείνοι που ε, δηλώνουν ότι έπεσαν θύματα διακρίσεων είναι πιο πιθανό να έχουν βιώσει σωματική και συναισθηματική βία. Αλλά υπάρχουν και άλλες μελέτες που αμφισβητούν τη σχέση μεταξύ είδους οικογένειας και νεανικού εγκλήματος. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μελέτη, η T-Side, η οποία ε, έγινε σε πολλές πόλεις της ε, βορειοανατολικής Αγγλίας το 2006 και δείχνει η μελέτη αυτή μια περιορισμένη σχέση μεταξύ είδους οικογένειας και αν ένα συγκεκριμένο άτομο νεαρό έχει υπάρξει παραβάτης ε, συχνά ή ποτέ. Υπάρχουν επίσης ε, μελέτες που ε, αμφισβητούν τη σχέση μεταξύ της σοβαρότητας και της συχνότητας των αδικημάτων. Επίσης υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η εστίαση δεν ε, ε, τοποθετείται σε παράγοντες κινδύνου όπως γονική ευθύνη. Επίσης καλό είναι να αναλυθεί η γειτονιά. Πολλές φορές γίνονται αδικήματα σε υποβαθμισμένες γειτονιές ενώ σε πιο πλούσιες περιοχές είναι λιγότερα συχνά τα αδικήματα ακόμα και αν υπάρχουν παρόμοιοι παράγοντες ε, επίπεδα κινδύνου το έγγραφο εργασίας νομίζω ότι πρέπει να τα λάβει όλα αυτά υπόψη ε, ως αποτελέσματα ερευνών. Δεύτερον, η εστίαση στην γονική ευθύνη δεν συνάδει, αν λάβουμε υπόψη μας, την αυτονομία των νέων. Δηλαδή την υποτιμά. Πολλές φορές και στις περισσότερες ε, ευρωπαϊκές χώρες Θεωρούμε ότι μπορούν να αναλάβουν ευθύνη για δικήματα και κάτω από τα, την ηλικία των 18. Από την άλλη, η ευθύνη των γονέων, και αν δούμε τη γονική ευθύνη, βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά ε, έχουν, αντιμετωπίζονται σ άτομα με καταλογισμό να διαπράξουν αδικήματα και κάτω των 18 ετών και από την άλλη οι γονείς ε, ε, θεωρούν ότι πηγαίνουν στο σχολείο και δεν ασκούν αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό ε, θα πρέπει να το δούμε μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας των νέων. Υπάρχει και μία μελέτη του 2000 των Γκόλτσον και Τζέιμισον ε, που εξέτασαν 49 νέους παραβάτες ε, και μόνο τρεις είπαν ότι θα μπορούσαν οι γονείς να έχουν προβεί αποτελεσματική διορθωτική δράση εις ό,τι αφορά την εγκληματική δραστηριότητα, η παραβατική δραστηριότητα. Θα ήθελα επίσης να επικεντρωθώ περισσότερο στη σχέση μεταξύ φύλου και ε, νεανικής παραβατικότητας. Ε, ήδη η κυρία Νόρντμπορκ το ανέφερε αυτό και νομίζω ότι είναι σημαντικό και το έγγραφο εργασίας ε, θεωρούμε ότι έχει μια μηχανιστική σχέση για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Γιατί η πολιτική για την ισότητα δεν πρέπει να στοχεύει στην ε, διασφάλιση του ελέγχου των γονέων πάνω στο παιδί. Ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι να ε, λύσουμε τις ιστορικές ανισότητες ανδρών και γυναικών. Επίσης, η προοπτική της γονικής ευθύνης στιγματίζει τις οικογένειες αφενός και την ποικιλομορφία τους, γιατί υπάρχουν οικογένειες που δεν ε, έχουν δύο γονείς, ούτε αποτελούνται από γονείς ή συντρόφους διαφορετικού φύλου. Αυτά θα μπορούσε κανείς να τα θεωρήσει παράγοντες κινδύνου, αλλά όπως είπα πιο πριν δεν υπάρχει διαπιστωμένη αιτιακή σχέση μεταξύ του ότι είναι μονογονική οικογένεια μια οικογένεια και το γεγονός ότι το παιδί που έβγαλε ε, ε, έχει παραβατικότητα. Επίσης ε, είναι σημαντικό να δούμε το ρόλο του άνδρα του... και το ρόλο που παίζει το πρότυπο του ανδρισμού στην ενική παραβατικότητα. Ε, έχει ασχοληθεί σε μια μελέτη, μια μελέτη με αυτό το θέμα από τον Οργανισμό Θεμελιωνόδων Δικαιωμάτων που δείχνει κάποια ε, αποτελέσματα ε, συνηγορούν υπέρ της σωματικής βίας κυρίως ε, από παιδιά που προβάλλουν τον ανδρισμό τους. Αν και παίζει λοιπόν ρόλο ο ανδρισμός στην ενική παραβατικότητα, ε, υπάρχουν και πολλές νεαρές κοπέλες που διαπράττουν παρόμοιες πράξεις. Αυτό φαίνεται σε άλλες έρευνες. Μια έρευνα, για παράδειγμα, του Πίτερσον το 2007 που δείχνει ότι 49 γυναίκες που έδωσαν συνέντευξη και είχαν διαπράξει κάποια βία η πράξη το προηγούμενο 12 μήνο πριν από την έρευνα, ε, το 61% Α, 49% γυναικών, 61% των ε, ανδρών, των νεαρών ανδρών είναι υψηλότερο το ποσοστό, αλλά βλέπουμε ότι είναι αρκετά σημαντικό, 49% και των νεαρών γυναικών που βιοπραγούν. Επίσης, ο ρόλος της ε, εκπαίδευσης, της παιδείας θα πρέπει να ε, τονιστεί περισσότερο στην έκθεση. Η γονική ευθύνη ε, βλέπετε μέσα από μια τιμωρητική προσέγγιση χωρίς να λαμβάνει υπόψη προληπτικά μέτρα για την ενική παραβατικότητα, όπου ένα από τα σημαντικότερα είναι η εκπαίδευση βέβαια, μέτρο πρόληψης. Θα πρέπει να υπάρξει εντονότερη εστίαση στην εκπαίδευση ως μέτρο πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας λοιπόν και Υπάρχει και το θέμα των μέτρων συμφιλίωσης συμβιβασμού που είναι σημαντικό μέτρο μεν. Είναι σημαντική αυτή η διαμεσολάβηση ε, που αναφέρθηκε και από τους άλλους εμπειρογνώμονες, αυτή η συνδιαλλαγή. Αλλά το σκεπτικό του μέτρου πίσω από αυτή τη συνδιαλλαγή, η συμφιλίωση, η συνδιαλλαγή, είναι να κατανείμει τις ε, οικογενειακές ευθύνες μεταξύ ανδρών και γυναικών ίσως χωρίς να δείχνει τόσο πολύ να επικεντρώνεται στις ιστορικές ανισότητες. Σε αυτό το τελευταίο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εστιαστούμε και όχι στην προληπτική και τιμωρητική προοπτική για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Θα ήθελα να τέλος να προτείνω και κάποιες πολιτικές δράσεις είναι πολύ πλευρό το θέμα της νεανικής παραβατικότητας, άρα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με διάφορες πολιτικές. Σίγουρα το πρώτο είναι οι πολιτικές που θα προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών και ειδικότερα σε αυτό το τομέα πολιτικής η εστίαση θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου. Εκεί πρέπει να δυναμώσουμε τις προσπάθειες, ιδιαίτερα μετά τον οδικό χάρτη 2006-2010 για την ισότητα ανδρών γυναικών. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση για την καταπολέμηση λοιπόν, ε, ε, στερεοτύπων φύλου και είναι θετική εδώ η έκθεση Φιγκερέιντο η οποία εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρώνεται πολύ στα στερεότυπα και την ανάγκη καταπολέμησης στερεοτύπων φύλου. Ένας άλλος τομέας πολιτικής, όπως προανέφερα, είναι σίγουρα η εκπαίδευση. Για παράδειγμα, σε αυτό το τομέα είναι σημαντικό, θεωρούμε, ε, να συμπεριληφθούν και σε αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης benchmarking σε σχέση με την εγκατάλειψη του σχολείου ε, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε και ε, σε αυτό το θέμα, να μην φεύγουν νωρίς από το σχολείο και στα πλαίσια των στόχων ήγιου 2020 2020 και οι προοπτικές φύλου θα πρέπει να ειδωθούν και σε αυτό το πρόβλημα ε, ως επιτοπλίστων τα αγόρια ε, έχουν διπλάσιο κίνδυνο και πιθανότητα να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο από ότι τα κορίτσια. Ένα άλλο τομέα πολιτικής που πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί είναι σημαντικό είναι η πολιτική GLS, το νέο Στοκχόλμη Στοκχόλμης 2010-2014 επικεντρώνεται πολύ σε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει ε, τις ριζοσπαστικές ε, στάσεις και τη βία. Θα υπάρξει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια στρατηγική αντιμετώπιση του ριζοσπαστισμού, ε, ραντικαλισμού και σε αυτό το τομέα της πολιτικής θα πρέπει να ενισχυθεί η εστίαση στην εκπαίδευση ως μέτρο πρόληψης και επίσης υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης διακρίσεων και κοινωνικών αποκλεισμών. Πρέπει να θεωρηθεί αυτό ένα από τα πιο σημαντικά ε, μέτρα πρόληψης του ριζοσπαστισμού των νέων. Τέλος, οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης, ε, οι πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας θα πρέπει να παίξουν ρόλο προληπτικό για την νεανική παραβατικότητα, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ε, αυτό το έτος είναι σημαντική ευκαιρία για μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές και γειτονιές, όπως είπα, γιατί υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ υποβαθμισμένων γειτονιών και ε, νεανικής παραβατικότητας. Κοινωνική ένταξη λοιπόν και μέτρα κατά της φτώχειας θα πρέπει να, να, είναι, να έχουν και γεωγραφική στόχευση για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στις υποβαθμισμένες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία, κυρία Περολίνη που συμβάλλατε στη συζήτησή μας και εσείς. Νομίζω ότι φωτίσαμε τις πλέον διαφορετικές πτυχές μέσα από τις ε, παρεμβάσεις και αυτό είναι σημαντική και πολύτιμη συμβολή για τις περαιτέρω διαβουλεύσεις μας. Ευχαριστώ θερμά και πάλι όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές και είμαι βέβαιη ότι θα ε, τεθούν και ερωτήσεις από τους παρευρισκομένους, ούτως ώστε να ε, πάμε σε περισσότερο βάθος σε αυτή την προβληματική. Εάν υπάρχει εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τώρα είναι η ώρα να λάβει το λόγο. Φαίνεται όμως ότι από την Κομισιόν δεν έχει έρθει κανείς. Τώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει κανείς. Εντάξει. Τότε το λόγο έχει η Επιτροπή, τα μέλη της αλλά και άλλοι σύνεδροι μπορούν να λάβουν το λόγο εάν έχουν να κάνουν ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες. Αρχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια. Να δώσω πρώτα το λόγο στην σκιώδη εισηγήτρια κυρία Σίμινσεν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, λυπούμε πολύ που καθυστέρησα να φτάσω. Άρχισε όμως το αεροπλάνο μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τον έγγραφο εργασία. Από ό,τι καταλαβαίνω πρόκειται απλά και μόνο για την απαρχή των εργασιών μας. Ω κοιότη εισηγήτρια στην ομάδα εργασία, ε, θέλω να συμφωνήσω με την εισηγήτρια που μιλά για την ενίσχυση του ρόλου τη οικογένεια για την καταπολέμηση της νεανικής παραβατικότητας. Ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε από ευρύτερο πρίσμα το όλο ζήτημα. Ε, υπάρχει και ένα οικονομικό ζήτημα το οποίο αναφέρεται, δηλαδή το επίπεδο, το βιωτικό της οικογένειας κτλ. Είναι καλή αυτή η προοπτική, είναι σωστή, δεν αρκεί όμως, διότι οι εγκληματικέ πράξει στι οποίε προβαίνουν οι νέοι μπορούν να σχετίζονται και με πολλέ άλλε πτυχέ και διαστάσει. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περιορίζουμε το πρίσμα αυτό, γιατί έτσι υπονομεύουμε τη σημασία του εγγράφου. Πράγματι, οι προβολείς πέφτουν κυρίως στην οικογένεια, αλλά όταν λέμε ότι η εγκληματικότητα η νεανική ε, σχετίζεται μόνο με μονογονεϊκές οικογένειες, αυτό δεν αληθεύει. Εάν ο πατέρας ε, χειροδική κατά της ε, συζύγου του ή των παιδιών του, περιμένουμε να μην μεταφερθεί η βία αυτή ε, και από τα παιδιά σε τρίτα άτομα. Το 50% των γάμων καταλήγουν σε διαζύγιο στην Ευρώπη και αυξάνονται τα ποσοστά. Εάν ε, όλοι, αν το περιβάλλον μιας τέτοιας οικογένειας ε, οδηγεί σε παιδιά βία, τότε το πρόβλημα δεν θα έχει ε, καμία διέξοδο και καμία λύση. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαθετήσουμε πολιτικές και να αλλάξουμε και την τροπία που έχουμε απέναντι στη βία. Δηλαδή, αν κατά κάποιο τρόπο δεχόμαστε κάποιες ε, παροιμίες που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες γλώσσες όπως τα πολωνικά ε, που λέει ότι όποιος αγαπάει παιδεύει κατά κάποιο τρόπο δηλαδή ότι ο άντρας που δέρνει τη γυναίκα του ουσιαστικά εκδηλώνει την αγάπη του. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την ισότητα των δύο φύλων για να μειώσουμε την ενική εγκληματικότητα, αλλά θα πρέπει να ε, προάγουμε, να προβάλλουμε και τα καλά πρότυπα και παραδείγματα. Θα πρέπει να βλέπουμε και κάποια ψυχοπαθολογικά προβλήματα, ε, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, γενετήσια, βία, σεξουαλική κακοποίηση κτλ. Ένα σημαντικό ποσοστό νεαρών εγκληματιών είναι παιδιά τα οποία έχουν νιώσει ε, ανεπιθύμητα, ε, δεν έχουν νιώσει αγάπη, ζουν μέσα σε ψυχρές οικογένειες χωρίς αγάπη. Ε, υπό αυτές τις συνθήκες η βία και η κλιματικότητα ίσως έρχονται και ως ε, φυσικές συνέπειες και για άτομα που μπορεί να ζουν απομονωμένα σε κάποιες χώρες κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να προάγουμε και τις μεθόδους αντισύλληψης, θα πρέπει να αποφεύγουμε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν απαραίτη, την απαραίτητη ενημέρωση για να μπορούν ε, να ε, κάνουν και άμβλωση ενδεχομένω, έκτρωση. Πάντως υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία γεννιούνται ε, λόγω ανεπιθύμητη εγκυμοσύνης. Υπάρχουν σε πολλές χώρες ε, αυστηροί νόμοι κατά των αμβλώσεων. και στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί νόμοι. 200 με 400 εκτρώσεις γίνονται νόμοι και 100.000 παράνομα. Το 1996 αποφάσισε το Συνταγματικό Δικαστήριο ότι είναι ε, αντίθετο με το Σύνταγμα, ε, κάτι που δεν ισχύει γιατί και σε άλλες ε, χώρες ισχύει ισχύουν ανάλογες διατάξεις στο Σύνταγμα. Υπάρχουν καθηγητές δικαίου, καθηγητές νομικής και δικαστές, πρόεδρες σταγματικών δικαστηρίων που όταν καταφέρονται κατά του δικαιώματος της άνδρας παραδείγματος χάρη, δημιουργούν κάποια άσχημα προηγούμενα. Η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη δεν είναι θετική. Επίσης η αγωγή στα σχολεία θα πρέπει να περιλαμβάνει ε, και τα θέματα της βίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστήσουμε περισσότερο την προσοχή και στην εκπαίδευση των ε, εκπαιδευτικών, των δασκάλων, που θα πρέπει να μπορούν και αυτοί να αντιδρούν σε φαινόμενα βίας ε, από μαθητές ή σπουδαστές. Και βέβαια η τιμωρία συμπεριφορών τέτοιου είδους ε, θα πρέπει να είναι αναπόφευκτη. Θα πρέπει τα παιδιά να σέβονται τη διαφορετικότητα, να σέβονται τις διαφορετικές συμπεριφορές. Έχουν αλλάξει βέβαια λίγο τα πράγματα, γιατί τα κορίτσια παραδείγματος ε, χάρη δεν έχουν μακριά μαλλιά, αλλά όταν ήμουν εγώ στο σχολείο τα αγόρια τράβαγαν τα μαλλιά των κοριτσιών. Ε, τώρα δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα βέβαια. Σίγουρα είναι διαφορετικά τα πράγματα μεταξύ, ανδρο... μεταξύ κοριτσιών και αγοριών. Η σεξουαλική δραστηριότητα ε, των κοριτσιών ε, ε, ενοχοποιείται κατά κάποιο τρόπο, όχι όμως των αγοριών όταν ε, παραδείγματο χάρη γίνονται βιασμοί λόγω και των κοινωνικών συνθήκων ε, οι γυναίκες δεν τις δηλώνουν, δεν τις καταγγέλουν ε, σε πολλές περιπτώσεις διότι είναι ταπεινωτικό το ότι υφίστανται ερωτήσεις του κατά πόσον φορούσαν πολύ κοντή φούστα η οποία μα προκάλεσε κτλ. Πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν ε, η ηλική κατάσταση στις οικογένειες, ε, ε, πρέπει να αλλάξει και το εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία. Αλλά θα πρέπει να καταπολεμηθεί γενικότερα κάθε μορφή ενδοικογενειακής βίας. Το έγγραφο τονίζει ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία ουσιαστικά να πω και τα αποκλειστικά στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει και αυτή το δικό της ρόλο, σεβόμενη με την αρχή της επικουρικότητας, αλλά σε κάποια κράτη-μέλη, λόγω του ότι πράγματι δεν υπάρχει διάκριση ε, μεταξύ κράτους και εκκλησίας, ή διότι υπάρχει πραγματική διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών, οι κυβερνήσει των κρατών αυτών δεν μπορούν να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά, τα προβλήματα αυτά, διότι δεν τα βλέπουν. Και έτσι επαφίενται, ε, μάλλον πολλές φορές ε, καταφεύγουν στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα στο πλαίσιο τη αρχή τη επικουρικότητα να βοηθήσει τα κράτη-μέλη εκείνα, την κυβερνήσει των οποίων δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, σωστά την ε, νεανική εγκληματικότητα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Εξετίμησα δεόντως αυτά τα οποία είπε στην αρχή της συζήτησης η κυρία Ζαμπόρσκα και η προσκεκλημένη μας. Να μου επιτρέψετε να κάνω κάποια σχόλια για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει και αυτό να αναζητήσει το τι μπορεί να γίνει. πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε σωστά ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου τους οποίους έχουμε μπροστά μας. Υπάρχουν ε, μελέτες, υπάρχουν έρευνες του ΟΗΕ, του ΟΣΑ για να δούμε ποια είναι τα βιώματα των ε, παιδιών, ποια είναι τα βιώματα των εφήβων και ποια είναι η τάση την οποία έχουν προς την εγκληματικότητα ή και ποια η ανοχή την οποία επιδεικνύουν σχετικά με την εγκληματικότητα. Εδώ έρχεται το θέμα του κοινωνικού περιβάλλοντος, το οποίο δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί, αυτό υπόθηκε προηγουμένως και συμφωνώ. Υπάρχει το θέμα της εκπαίδευσης. Πολλές ε, έρευνες δείχνουν ότι η σχέση ανάμεσα στην εγκατάλειψη του σχολείου και στις αντικοινωνικές συμπεριφορές είναι δεδομένη. Είναι αποδεδειγμένη, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ίσως μέχρι τώρα λίγο να λείπει από αυτή την συζήτηση είναι το λεγόμενο peer education, δηλαδή τα πρότυπα τα οποία μπορεί να έχουν τα παιδιά. Όταν υπάρχουν αντικοινωνικές ή μη κοινωνικές εν πάση περιπτώσει συμπεριφορές, η μη κοινωνικες σε παση περιπτωσει συμπεριφορες η κοινωνια των πολιτών, οι οργανώσεις που φροντίζουν τα παιδιά, οι αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να βοηθήσουν. Μπορεί να υπάρξει μια ισχυρή υποστήριξη προς κάποιες δραστηριότητες οι οποίες ε, ε, ασκούν θετική επίδραση στα παιδιά. Να προωθηθεί γενικά η κουλτούρα της συνεννόησης, της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και αυτό ίσως μπορέσει να μας βοηθήσει να δούμε ε, ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα παρέμβουμε. Μας λέγει η συγγήτρια με το θέμα του τι θα πρέπει να κάνουν οι οικογένειες. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να παρανοηθεί γιατί είναι εύκολο να κατηγορήσει κανείς κάποιες οικογένειες για τη συμπεριφορά τους, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε παρά να πάρουμε υπόψη μας το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και κινούνται οι οικογένειες. Και υπάρχουν και πολλές μορφές οικογένειας, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες. Θα πρέπει λοιπόν να μην αγνοήσουμε την οικογένεια, δεν είναι ιδεολογικό το θέμα, το θέμα είναι ότι θέλει όμως πάρα πολύ προσεκτική παρουσίαση. Και θα πρέπει χωρίς να στιγματίσουμε κάποιες μορφές οικογένειας όπως τη μονογονεϊκή οικογένεια και οι μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνονται συνεχώς και αυξάνονται και τα παιδιά λοιπόν που ζουν με έναν γονιό μόνο θα πρέπει να μην είμαστε ουδέτεροι σε επίπεδο κοινωνικών πολιτικών και γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα δικαιοδοσίας εδώ, ε, τοπικό και εθνικό, να πούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σε επίπεδο γενεών και σε επίπεδο ευελιξίας ωραρίου εργασίας για τις γυναίκες και για τους αρχηγούς των οικογενειών και φυσικά αυτό θα πρέπει να αφορά και τις μονογονικές οικογένειες. Αναφερθήκαμε στην εγκληματικότητα με πολύ γενικό τρόπο. Ίσως θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο το αν μπορεί να υπάρξει ένας ορισμός κάπως πιο συγκεκριμένος. Γιατί έχουμε από τη μία την οργανωμένη αν θέλετε εγκληματικότητα από την άλλη έχουμε ένα διαφορετικό φαινόμενο, το bullism όπως λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή την άσκηση άτυπης βίας ε, σε καθημερινή βάση στα σχολεία κτλ. Εκεί πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις σε επίπεδο χρηστών πρακτικών θα έλεγα, έτσι ώστε αυτό το bullism που είναι η βία στα σχολεία ή στους χώρους τους κοινωνικούς των νέων έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει, ακόμα και σε οικογενειακό περιβάλλον και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Η Ελίζα Μάνα έχει δίκιο ότι το πρότυπο το οποίο εμείς μεταφέρουμε μέσα από την ενημέρωση στην ουσία είναι ένα πρότυπο το οποίο πηγαίνει τη γυναίκα πίσω και είναι ο προθάλαμος της άσκησης βίας εις βάρος της γυναίκας από πλευράς των ανδρών αλλά όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Να ευχαριστήσω και εγώ τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι πήραν το λόγο σήμερα.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 την ποιότητα των παρεμβάσεών τους, να ευχαριστήσω και την κυρία Μάνα για την παρουσίαση την οποία έκανε για την κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να δει τη γυναίκα και να κρίνει τη γυναίκα μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Και εγώ συμφωνώ με την κυρία Μάνα όταν ταξιδεύω στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω διαφημίσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα ακραίες εις βάρος της γυναίκας. Και ακόμα και ένα λάστιχο αυτοκινήτου να διαφημίζεται πάντα υπάρχει μια ημίγυμνη γυναίκα ακριβώς δίπλα. Ε, intervento e quindi spunto del, ε, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Περολίνη όταν αναφέρθηκε στην ευθύνη των γυναικών, στην ευθύνη την οποία μπορεί να έχουν γενικότερα οι νέοι και στον έλεγχο των συμπεριφορών τους. Όπως είπε ήδη η κυρία Κώστα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Και εδώ έρχονται οι προτάσεις και τα σχόλια τα οποία έχει ήδη κάνει η κυρία Ζαμπόρσκα. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες διευκρινήσεις για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει τις πολιτικές ισότητας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στα πλαίσια της καταπολέμησης και της καταπολέμησης της παιδικής και νεανικής εγκληματικότητας πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό το ταχύτερο δυνατόν. Εν περιπτώσει μέχρι τώρα νιώθω μια κάποια απογοήτευση από τις προτάσεις που έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά να ευχαριστήσω την κυρία Ζαμπόρσκα για την προσπάθεια την οποία έκανε και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, τη συνεισηγήτρια ε, ή τη σκιώδη μάλλον εισηγήτρια για αυτά τα οποία μας είπε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματέρα. είπα να εκφράσω και εγώ κάποιες απόψεις μου. Καταρχήν, η Επιτροπή μας καλείται να λάβει υπόψη της την ισότητα ευκαιριών σε όλες τις πολιτικές, γιατί έτσι θα συμβάλλουμε ώστε να περάσει το μήνυμα ε, ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον αποκλεισμό την εγκληματικότητα μέσα από πολιτικές. Αυτή είναι η δική μας συμβολή στην ευρύτερη συζήτηση. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες γιατί είμαι πεπισμένη ότι εδώ ακούσαμε πολύτιμα και σημαντικά πράγματα. Εγώ παρακολουθώντας προσεκτικά τους εμπειρογνώμονες έμαθα πολλά. Προσέθεσα γνώσεις και νομίζω ότι μπορώ στο έργο μου στο μέλλον να αξιοποιήσω πλήρως αυτά που μας είπατε. Είναι σημαντικό και για την εισηγήτρια ε, το ότι ακούσαμε τους εμπειρογνώμονες. Τώρα στο έγγραφο εργασίας ε, σε μεγάλο βαθμό ε, η εστίαση βρίσκεται στην οικογένεια. Νομίζω ότι συχνά αυτό που βλέπουμε είναι η κοινωνική πραγματικότητα διαφορετικών ομάδων. Γιατί υπάρχουν μελέτες που συμπεραίνουν ότι ο κίνδυνος ε, της εγκληματικότητας αυξάνεται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Φαντάζεστε τι προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει μια οικογένεια ανάλογα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Αν ζει μέσα σε φτώχεια, αν δεν μπορεί να προσβλέπει με εμπιστοσύνη το μέλλον, αν οι γονείς αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μπούμε στη θέση τους και να δούμε πώς ένας γονιός μπορεί να δώσει εμπιστοσύνη στο μέλλον στο παιδί του όταν ζει ή στην κοινωνία, όταν ζει μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Είναι λοιπόν απόλυτα σημαντικό να αυξήσουμε τις ευκαιρίες για όλους και να μην αφήσουμε ανθρώπους να νιώθουν ότι έχουν αποκλειστεί, έχουν περιθωριοποιηθεί, αλλά όχι ότι είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και πρέπει να ε, εστιάσουμε στους μηχανισμούς στήριξης που υπάρχουν για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, ε, διαφοροποιούμε λίγο ως προς το θέμα της ακέραιης ή της ατελούς οικογένειας, της ελιπούς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι όροι. Πώς θα ορίσουμε την οικογένεια που θα έχουμε. Μιλάμε για μονο, είτε μιλάμε για γονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες όπου και οι δύο γονείς είναι του ιδίου φίλου, οι οικογένειες όπου υπάρχουν άνδρας γυναίκα στην οικογένεια. Όλες οι οικογένειες όμως μπορούν να έχουν τις ίδιες αξίες και είναι σημαντικό εμείς να αναγνωρίσουμε όλες τις μορφές αυτές της οικογένειας γιατί όλα ασκούν τον υποστηρικτικό τους ρόλο. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί αυτή τη δουλειά και θέλω τέλος να κάνω μια ερώτηση στους εμπειρογνώμονές μας. Πολύ συχνά όταν ακούμε περιγραφές για αυξημένο κίνδυνο εγκληματικότητας και όταν ζούμε σε ε, οικογένειες χωρισμένες, ε, διαζευγμένες κλπ. Θα πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί πριν από το διαζύγιο, γιατί το παιδί συχνά έχει γίνει μάρτυρας βίαιων καταστάσεων, έχει βιώσει δυσλειτουργικές σχέσεις. Δεν είναι αυτό καθοριστικό ή σε ποιο βαθμό είναι καθοριστικό για το μέλλον του παιδιού. Δεν είναι αυτό σημαντικό και όχι μόνο η ζωή του παιδιού μετά το διαζύγιο με τον ένα γονέα. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό και τη σημασία αυτών των καταστάσεων. Δεν έχω άλλον γραμμένο στον κατάλογό μου για να λάβει το λόγο, οπότε προτείνω τώρα να δώσουμε πάλι το λόγο στους τρεις προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν στα σχόλια και τις ερωτήσεις και να προσθέσουν και άλλες παρατηρήσεις αν θέλουν. Πρώτα η κυρία Νόρντμπορκ. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία. Ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικές συνεισφορές από τους ε, συναδέλφους μου, εδώ τους διπλανούς εμπειρογνώμονες, αλλά και από άλλους που έλαβαν το λόγο. Έτσι για να τα κάνω πιο απλά τα πράγματα θα απαντήσω πρώτα στο τελευταίο. Αν γνωρίζουμε, ο υψηλός κίνδυνος εγκληματικότητας εξαρτάται από το ότι το παιδί ζει σε μονογονική οικογένεια ή από το τι έχει συμβεί πριν. Εγώ νομίζω το είχα πει και πριν. Ε, είναι εύκολο το ερώτημα, δύσκολη απάντηση όμως. Έχει γίνει πολλή έρευνα. Η οποία βασίζεται σε στατιστικούς παράγοντες. Ίσως το υπόβαθρο είναι πράγματι ότι κάποιο παιδί που έχει εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά ζει σε μονογονεϊκή οικογένεια, σε τέτοιο περιβάλλον. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, Πολύ λίγη έρευνα έχει γίνει με συνεντεύξεις των ατόμων και σύνδεση, διασύνδεση με το περιβάλλον. Δηλαδή δεν είναι στατιστικός ε, ασφαλή τα συμπεράσματα για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η κατάσταση. Υπάρχει κάποια έρευνα επίσης που έχει γίνει η οποία παρακολουθεί εκ του σε αυτά τα νερά άτομα με συνεχείς συνεντεύξεις και εκεί είναι προφανές ότι Ο παράγοντας κινδύνου και αυτό που έχει βλάψει πραγματικά αυτά τα παιδιά είναι η βία. Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε κάτι σε αυτόν τον κατάλογο και αυτό θα ήταν να γίνει περισσότερη έρευνα και περισσότερη έρευνα βασισμένη ε, στη διάσταση του φύλου. Και επίσης θα πρέπει να γίνουν και μελέτες πάνω στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα και στην πρακτική τους εφαρμογή. κυρία Κώστα νομίζω ρώτησε κάτι. Αν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο και να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αυτό έχει σχέση και με το τι ε, εννοούμε όταν λέμε βία, όταν λέμε εγκλήματα ή εγκληματικές πράξεις. Εγώ περιλαμβάνω τα πάντα εδώ, όλες τις μορφές. Νομίζω ότι και στην Εύνα υπάρχει τάση όταν λέμε βία να εννοούμε την σωματική βία, την οικογενειακή βία, τη σεξουαλική βία, μέχρι και το θάνατο, τη δολοφονία, που και αυτό μπορεί να συμβεί φυσικά. Νομίζω επίσης ότι αρχίζουμε πια όλο και περισσότερο να ε, κοιτούμε όλους τους τύπους. Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή αλλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάποια μικρότερα πράγματα. Δηλαδή κάποια αστεία που τα δεχόμαστε, ότι λέμε εντάξει έτσι φέρονται τα γόρια. Αλλά αυτό αν το αφήσουμε να αναπτυχθεί επιδεινώνεται. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιο θύμα εκφοβισμού, bullying, επίσης θα πρέπει να το προσέξουμε. Και τα θύματα δηλαδή πρέπει να τα προσέξουμε για να εμποδίσουμε το να οδηγηθούν λόγω της αγανάκτησης, της οργής που νιώθουν, του άγχους τους, ε, να στραφούν και αυτά στη βία, σε βίες ενέργειες. Υπάρχει μεγάλη σχέση το θύμα να γίνει θήτης κάποια στιγμή. Νομίζω θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επανέλθω σε αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως μετά από το εξαιρετικό ε, έγγραφο το οποίο συνέταξε η κυρία Ζαμπόσκα. Ξεκινώ από το ερώτημα το οποίο θέσατε. Σημερίζομαι το ότι θα πρέπει να υπάρξει πολύ περισσότερη έρευνα σε σχέση ε, με τη βία και την οικογένεια. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και στα οποία μπορούμε να αναφερθούν μας δίνουν την δυνατότητα θα έλεγα να πούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος να είναι κανείς μάρτυρας σκηνών βία στην οικογένεια και με συστηματικά βίαιες συμπεριφορές στα πλαίσια της υιοθέτηση ενός βίαιου προτύπου καθημερινής διαβίωσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Φυσικά και οι μονογονεϊκές οικογένειες πολλές φορές ε, βλέπουν να δημιουργούνται οικογένειες, προβλήματα και τέτοια φαινόμενα. Αλλά από ό,τι γνωρίζουμε από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, οι σκηνές βίας ας πούμε της τηλεόρασης και οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας ε, των γυναικών γενικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο συστηματικό και επηρεάζει τα παιδιά. Το θέμα του ρόλου της τηλεόρασης και των μέσων ενημέρωσης γενικά πάνω στο συγκεκριμένο αυτό θέμα. Θα ήθελα να σας πω, χωρίς να υπάρξει ιδιαίτερα φόβος διάψευσης, ότι τα επιστημονικά στοιχεία ε, στο συγκεκριμένο τομέα είναι επιβλητική. Η πρώτη μελέτη η οποία απέδειξε τον συσχετισμό ανάμεσα στην τηλεοπτική βία και την συμπεριφορά την βίαιη των παιδιών ε, έχει γραφτεί από το 1957 το London School of Economics. Λεγόταν η μελέτη αυτή Television and the Child. Από τότε στις Ηνωμένε Πολιτείε στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις υπόλοιπες χώρες και αναφέρομαι εδώ στην επιστημονική παραγωγή στον Καναδά και την Αυστραλία έχουν αποδείξει συστηματικά θα έλεγα την σαφέστατη σχέση ανάμεσα στην τηλεοπτική παρουσίαση της βίας και τις βίαιες συμπεριφορές των νέων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει φαντάζομαι και γι' αυτό είμαι στη διάθεσή σας για να σας δώσω ακριβώς αυτήν την επιστημονική βιβλιογραφία την οποία θεωρώ όπως είπα επιβλητική. Άλλωστε το Τσένσις έχει επιφορτιστεί από την ανεξάρτητη αρχή της Ιταλίας για τη βία να ε, διατυπώσει και μία λευκή βίβλο για την βία στην τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα. Συνεπώς, η σχέση τηλεόρασης και ε, παιδιών στον τομέα της η συμπεριφοράς είναι δεδομένη. Υπάρχουν δέκα θα έλεγα βιβλία τα οποία επιβεβαιώνουν τη σχέση αυτή και ένα κάθε φορά το οποίο την αμφισβητεί. Λοιπόν, το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αντιπαρατεθούμε σε αυτήν την επιρροή. Να μου επιτρέψετε να επανέλθω αυτό στο λεγόμενο family mainstreaming. Νομίζω ότι είναι μια σωστή ε, κατεύθυνση. Να πούμε δηλαδή ότι το οικογενειακό πλαίσιο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλες τις πολιτικές τις οποίες ακολουθούμε. Στο έγγραφο ε, περιλαμβάνεται και μια Ιταλική εμπειρία θετική της πόλης Πιστόια Μια εμπειρία η οποία θα μπορούσε θα έλεγα να χαρακτηριστεί σαν μία από τις α, ε, α, ε, πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι οικογένειες να μην νιώθουν απομονωμένες, να νιώθουν ότι καλύπτονται οι ανάγκες τους τοπικά, να νιώθουν ότι είναι ικανές να διαχειριστούν τις εσωτερικές τους αντιθέσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει σε μικρό, ε, θα έλεγα, σε μικρή κλίμακα να υπάρξουν υπηρεσίες οικογενειακού τύπου στα πλαίσια των οποίων να υπάρχει δυνατότητα εκτόνωσης των αντιπαραθέσεων μεταξύ των γενεών και αντιμετώπισης των προβλημάτων των διαφόρων γενεών και των πόρων θα έλεγα και των συνεισφορών που μπορεί μία γενεά να προσφέρει στην άλλη. Υπάρχει εδώ μία θα έλεγα επικουρική σχέση ανάμεσα στις γενναίες με την βοήθεια μιας ειδική υπηρεσίας βέβαια γιατί πολλές φορές ε, δεν υπάρχει ανάγκη να γίνουν τεράστιες προσπάθειες ε, ε, για να ξεκινήσει μια διαδικασία συμφιλίωσης και συνεννόησης, μια μορφή counseling, συμβουλών. Λοιπόν, η τηλεόραση μπορεί να λειτουργήσει και προς την κατεύθυνση αυτή μέσω τηλεοπτικών προγραμμάτων που να ευνοούν την ισότητα των φύλων. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Περολίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στα όσα είπαν οι ευρωβουλευτές Κώστα και Ματέρα. Ο εκφοβισμός, το μπούλισμ, είναι μια μορφή βίας πράγματι και θεωρείται και από την έρευνα ως μορφή βίας και σε παλιότερες έρευνες θεωρείται μορφή βίας. Σύμφωνα με τον, την νομοθεσία για την ισότητα είναι μορφή διακρίσεων ο εκφοβισμός, μπούλισμ. Το πρόβλημα είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυστυχώς, παρόλο που πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ε, δεν υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή που παρέχει προστασία στην εκπαίδευση κατά ε, σε περίπτωση τέτοιων ε, αδικημάτων. Δεν υφίσταται σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το μπούλισμ είναι μια μορφή παρενόχλησης αλλά και διακρίσεων με βάση τον νόμο περί ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν την χάνει προστασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εγκρίνουν νομοθεσία ε, για την ισότητα που θα καλύπτει και τις διακρίσεις ε, για λόγους φύλου κλπ. Αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα νομοθετικό κενό το οποίο οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πιστεύουν ότι πρέπει να καλυφθεί. Επίσης στην ομιλία μου μίλησα για την συνέχιση της στρατηγικής οδικού χάρτη για την ισότητα ανδρών γυναικών. Ήδη ανέφερα τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ νεανικών εγκλημάτων των νέων ε, προτύπων ανδρισμού και άλλων στερεοτύπων που υπάρχουν και τα είπαν οι συνάδελφοι και στερεότυπα ε, που προβάλλονται από τα ΜΜΕ και συμβάλλουν στην ένικη εγκληματικότητα. Οπότε θα πρέπει να δούμε την συνέχιση της στρατηγικής μας για την καταπολέμηση αυτών των στερεοτύπων και στην εκπαίδευση και αν και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση, στον τομέα της παιδείας είναι περιορισμένες, όμως ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα στερεότυπα των φύλων στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων. Αυτό είναι κατεπήγον. Και ο δικός χάρτης, η συνέχιση της στρατηγικής, είναι ευρωπαϊκή πολιτική και με κάθε σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας βέβαια και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα καταπολεμούν στον τομέα της εκπαίδευσης τα στερεότυπα των φύλων. Επίσης, υπάρχει η βία μέσα στις οικογένειες, ενδοοικογενειακή βία. Πολύ σημαντικό και αυτό γιατί δείχνει ότι η οικογένεια αυτή καθ' αυτή δεν είναι μια ιερή κοινωνική δομή, ένα, αλλά ε, μια δομή, ένα μόρφωμα που έχει ελλείψεις. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτή την προοπτική να την συνδέσουμε με τις πολιτικές ε, κατά της βίας σε βάρος γυναικών. Για παράδειγμα, σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης Υπάρχει ένα σχέδιο σύμβασης για τη βία κατά των γυναικών και σε αυτό το πλαίσιο ίσως μπορούν να προβλεφθούν μηχανισμοί προστασίας ε, και των έμεσων θυμάτων της βίας ε, όπως τα παιδιά μέσα σε αυτή την βία οικογένεια. Και το ίδιο ισχύει ίσως και για το πλαίσιο σύμβασης ε, για την ε, καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών. Στα πλαίσια αυτής της νέας πολιτικής και στρατηγικής θα πρέπει να δούμε και τον αντίκτυπο στα παιδιά της βίας μέσα στις οικογένειες αυτές. Varmt tack till Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εμπειρογνώμονες και τώρα η κυρία Άννα Ζαμπόρσκα, η συγγήτριά μας για τις καταληκτικές της παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κρίμα που έχουμε τόσο λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Από ό,τι κατάλαβα, Υπάρχουν πολλοί εδώ από το ευρύ κοινό, από μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίοι θα ήθελαν να λάβουν το λόγο στη συζήτηση. Από ό,τι φαίνεται όμω δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μα. Παρ' όλα αυτά, να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχάς ε, και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εμπειρογνώμονες και τους συναδέλφους ε, που παρέστησαν σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι ό,τι ακούσαμε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα ε, για να συνεχίσω την επεξεργασία αυτής της έκθεσης. Καταρχάς, ε, να αναφέρω ένα ζήτημα αρχής. Δέχομαι ότι η νεανική παραβατικότητα ως έννοια είναι ιδιαίτερα ευρεία. Υπάρχουν πολλά αίτια και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και πολλές ε, δυνητικές λύσεις. Όλο το ζήτημα θα πρέπει να ειδωθεί σφαιρικά Κάθε έκθεση όμως η οποία συντάσσεται, εάν αντιμετωπίζει τόσο σφαιρικά το πρόβλημα, δεν θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Θα τονίζει τις διάφορες πτυχές του, αλλά δεν θα μπορεί να προτείνει λύσεις. Όπως είπα, το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση για το ρόλο των γυναικών, της οικογένειας και της κοινωνίας για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. Αυτό σημαίνει ότι ήδη ένας τομέας έχει αντιμετωπιστεί. Στη δική μου έκθεση, στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, στόχος μου ήταν να τονίσω τις πολιτικές ε, της ισότητας ευκαιριών που θα δώσουν σε άνδρες και γυναίκες τη δυνατότητα να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την καταπολέμηση της νεανικής παραβατικότητας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Σφένσον, κυρία Πρόεδρε, που τονίσατε τις πολιτικές αυτές ε, της ισότητας ευκαιριών και τη σημασία που έχουν. Το έγγραφο εργασίας αναφέρεται ρητός στο ότι τέτοιου είδους πολιτικές που είναι πρόθυμες ε, να εκπονήσουν ε, και οι εθνικές ε, νομοθεσίες και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν να εναρμονίσουμε και να βελτιώσουμε το έργο το οποίο γίνεται από άνδρες και γυναίκες μέσα στην οικογένεια, για να καταπολεμηθεί έτσι τον ενικό, η νεανική εγκληματικότητα. Είναι κρίμα, κατά την άποψή μου, που σε αυτές τις παρεμβάσεις ασχοληθήκαμε με πολλές άλλες ε, πτυχές, αλλά όχι τόσο με τις πολιτικές της ισότητας ευκαιριών. Είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας κάθε είδους έρευνα. Υπάρχουν μεμονωμένες μελέτες που έχουν διεξαχθεί από εμπειρογνώμονες ή από μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή από ιδρύματα. Αν όμως διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο εργασίας μου, θα διαπιστώσετε ότι ίσως να είναι ιδιαίτερα υποκειμενικές αυτές οι μελέτες. Είπε ο κύριος Περολίνο ότι υπάρχουν και άλλες μελέτες. Με τα χαράς να αναφέρω όλες αυτές τις μελέτες και έρευνες, αλλά ο στόχος μου ήταν κυρίως να επικεντρωθώ σε έρευνες από πανεπιστήμια που υπό, από ευρωπαϊκά ιδρύματα, που ήταν κάποια σημεία αναφοράς για εμάς. Εγώ δεν έχω αναφέρει παρά μόνο τις αντικειμενικές και όχι υποκειμενικές μελέτες που μπορεί να επηρεάζονταν από συγκεκριμένη ιδεολογία. Ο κύριος Περολίνη είπε ότι υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της ε, γονικής ε, φροντίδας και της αυτονομίας. Χαίρομαι που το αναφέρατε αυτό, γιατί όλο και περισσότερο θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράδοξο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός, προσπαθούμε να ιδιωτικοποιήσουμε όλες τις υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις, τα διάφορα εγχειρήματα και από την άλλη πλευρά κρατικοποιούμε την ιδιωτική ζωή. Εγώ είμαι αυτή η οποία θα ήθελα να υποστηρίξω την αυτονομία της οικογένειας και της ιδιωτικής ζωής, αλλά βέβαια στο ε, σχετικό πλαίσιο. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά πρέπει να υπάρχει και αυτονομία. Δεν είμαι σύμφωνη με τις ε, κυρίαρχες τάσεις. Ακούσαμε επίσης να γίνεται λόγος για διάφορα είδη οικογενειών. Θέλω να πω όμως ότι αντικείμενο της έκθεσής μου δεν είναι η οικογένεια. Δεν είχα ως στόχο να επιχειρηματολογήσω ποια μορφή οικογένεια είναι η λιγότερο περισσότερο κατάλληλη για την καταπολέμηση της νεανικής παραβατικότητας. Αυτό το οποίο προσπαθούσα να τονίσω και να, στο οποίο προσπαθούσα να εστιάσω ήταν η οικονομική προσέγγιση. Θέλω να δώσω έμφαση εκεί. Θέλω να τονίσω το κόστος. για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Δηλαδή, ε, υιοθέτησα μια ηθικώς ουδέτερη προσέγγιση. Ήθελα να αναφερθώ σε ε, γεγονότα και στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. σίγουρα εντάσσεται όλα αυτά στο γενικότερο πλαίσιο της νεανικής εγκληματικότητας. Ήθελα όμως να αναφερθώ και στην ενδοοικογενειακή βία. Ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλοι είμαστε αντίθετοι στη βία μέσα στην οικογένεια. Είμαι πεπισμένη ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το ζήτημα έχει να κάνει με παραδείγματα, με το ρόλο του πατέρα, αν είναι βίος απέναντι στη σύζυγό του. Είναι ένα κακό παράδειγμα, αλλά μιλάω και για τα παιδιά. Τα παιδιά γίνονται όλο και πιο βία απέναντι στους γονείς τους. Πρέπει να τονίσουμε και την ανάγκη σεβασμού των γονιών από τα παιδιά. Το Συμβούλιο της Ευρώπης θα ψηφίσει ένα ψήφισμα για κάποια σεξιστικά στερεότυπα γυναικεία συγκεκριμένα στερεότυπα στην ε, Ευρώπη ή στα μέσα ενημέρωση, συγγνώμη. Η Ταλίδα γνωμη η μίλησε διαμακρών για την προβολή της γυναίκας από τα μίντια ως ενός σεξουαλικού αντικειμένου. Και όχι ως μητέρας, δεν προβάλλει τη γυναίκα ως μητέρα, αλλά ως αντικείμενο. Αν θέλουμε λοιπόν να αλλάξει αυτό, δεν θα πρέπει να εγκρίνουμε εκθέσει οι οποίε παρουσιάζουν την εικόνα τη μητέρα ω ένα σεξιστικό στερεότυπο. Κάποιες φορές ε, μπορούμε να, μπορεί να παρισφρήσουν λάθη έγγραφα τα οποία εγκρίνουμε και αυτά να επηρεάσουν ε, τους πολίτες, τους νέους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και σίγουρα προσβλέπω και σε μελλοντική μας συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχαριστώ και τους φιλοξενουμένους μας που ε, πήραν μέρος στη συζήτηση και μας βοήθησαν ιδιαίτερα. Θα συνεχίσουμε στην ημερήσια διάταξη. Ας προσπαθήσουμε τώρα να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Καλώς. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για την κοινωνική ένταξη των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες. Αυτή είναι μία έκθεση για την οποία οργανώσαμε τον μήνα Απρίλιο και μία ακρόαση. Τη συζητήσαμε στις 3 Μαΐου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Αντωνία Παρβάνοβα και τις δύο το λόγο αν θέλει να πει κάτι, να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Έχετε το λόγο κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους σκιώδεις συζητητές και τις πολιτικές ομάδες που με βοήθησαν σε αυτήν τη δύσκολη γενικά ευαίσθητη έκθεση. Έγινε μια μακρά συζήτηση που δεν αφορά μόνο τις δικές μας πολιτικές ομάδες, αλλά γενικότερα το θέμα αυτό και την κοινωνία. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες Όλες οι τροπολογίες ήταν συμβατές με τη φιλοσοφία της έκθεσης. Νομίζω ότι υπάρχει ένα περιβάλλον εργασίας ιδιαίτερα θετικό. Προσπαθήσαμε τις τροπολογίες αυτές να τις εντάξουμε στο κείμενο. Άκουσα τις παρατηρήσεις και των συνεισηγητών, των σκιωδών εισηγητών μάλλον. Οι περισσότερες επαναλαμβάνω από τις προτάσεις τροπολογιών οι οποίες ήλθαν από τους συναδέλφους ε, θα γίνουν δεκτές. Ελπίζω λοιπόν με τη θετική σας ψήφο να έχουμε μια ευκαιρία για την Επιτροπή μας να ακουστεί στην Ολομέλεια και να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Παρβάνοβα. Ήταν πολύ προσεκτική η δουλειά την οποία κάνατε. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε πλέον στην ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 60. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 61. Υπέρ. Κατά Αποχές. Κανείς δεν είναι κατά. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 4. Ο κύριος Σοβά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω μια προφορική τροπολογία να αναφερθώ στο θέμα της προστασίας των δεδομένων από τις εθνικές υπηρεσίες γιατί το θέμα των πληροφοριών που άπλονται της εθνότητας ε, ή της εθνοτικής μειονότητας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να, ε, ε, αυτό να λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια των εθνικών νομοθετικών ενέργειων. λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με τους κανόνες για την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Να αλλάξουμε τη φάση αυτή και να πούμε σύμφωνα με τους κανόνες των διαφόρων κρατών μελών για την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Υπάρχει αντίρρηση για αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ της 4. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Επανερχόμεθα τώρα στην 62. Ζητήθηκε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 62. Άρχεται η ψηφοφορία. 62. Τέλος. Απερίφθη. 10 ψήφισαν υπέρ, 20 κατά και απερίφθη. Στη συμβιβαστική 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 70, όχι, θα την ψηφίσουμε μετά. Η συμβιβαστική 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 7. Με μια προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 86. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 86. Ψηφίζεται. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν ε, έναν επιπλέον ψηφίζοντα. Η κυρία Πλάμπα πέσυρε την κάρτα της. Πέρας της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε εκ νέου για την 86. Πάντα ένας επιπλέον ψηφίζει από πλευράς των σοσιαλιστών. Ψηφίζουμε ξανά λοιπόν για την 86. Πέρας της ψηφοφορίας. 16 υπέρ 15 κατά. Τώρα 87 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 92. Με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 93, και 101 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε μαζί για τις τρεις ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 113. Ψηφίζουμε. Πέρα στη ψηφοφορία. Απερίφθη. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 71. Και εδώ υπάρχει προφορική τροπολογία για το δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές Απερίφθει. Εκατόν υπέρ. Κατά. Αποχές. απερίφθεια. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 135 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Το δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Συνεπώς. Περνάμε στο 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ελέγχουμε την 134. Vote Απερίφθηκε η 134. Πηγαίνουμε στην 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 140 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 139 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 143. Διακόπτη η πρόεδρος. Επανέρχομαι 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Πηγαίνουμε στην 147 και 148 που είναι ταυτόσιμες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 24. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 24. Απερίφθη. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α, Για την 27 έλεγχος ψηφίζουμε closed and it's rejected. Απερίφθη. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 39. Τέλος της ψηφοφορίας απερίφθη. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 31 υπέρ. Συγγνώμη, 32. 32 και 33 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Α, έλεγχος πάλι για την 32 και 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχει γίνει δεκτή. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 37 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 38 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Σαράντα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 41 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 43 και 44 ταυτόσιμες. Α, έχουν καταπέσει έτσι και αλλιώ πηγαίνουμε στη συμβιβαστική. Α, για μια στιγμή. 45 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα περνάμε στη συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 56 υπέρ. Όχι. Ψηφίζουμε ξανά. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 57 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 59 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τέλος, η 3 υπέρ, κατά, δεκτή. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πάντα οι σοσιαλιστές είναι ένας περισσότεροι. Συγχαρητήρια κυρία Παρβάνοβα. 28 υπέρ, κανείς κατά 11 αποχές. Ευχαριστούμε κυρία Παρβάνοβα, συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες και Περνάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας μιας νέας βιώσιμης οικονομίας είναι γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Απασχόλησης. Είχαμε σχετική συζήτηση στις 3 Μαΐου και η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ήταν η 11η Μαΐου, 44 τροπολογίες υπευλήθησαν και η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι η κυρία Τόμψεν. Έχετε το λόγο για τυχόν σχόλια πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι μια έκθεση η ονομοδότηση επί εκθέσεως για την ανάπτυξη δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας σε μια νέα πράσινη οικονομία. Θα επενδύσουμε στο μέλλον σε αυτήν. Δεν μπόρεσα να καταθέσω συμβιβαστικές τροπολογίες, γιατί οι τροπολογίες που κατετέθησαν αφορούν ολόκληρη σειρά διαφορετικών θεμάτων και γι' αυτό δεν είχαμε συμβιβαστικές. Όχι επειδή διαφωνούσαμε όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τόμσεν. Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 12 σε τρία μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και το τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος στο τρίτο το, μέρος της τροπολογίας 12 άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι το ίδιο, ε, μία ψήφος παραπάνω στους σοσιαλδημοκράτες. Πέρασε της ψηφοφορίας, εντάξει είναι τώρα. Δεκτό 18 υπέρ και 13 κατά. Δεκτό πάντως. Προχωρούμε. Τροπολογία 14 καταπίπτει. 15 σε δύο μέρη. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Καταπίπτει. Θα πάμε στην τροπολογία 16. Υπέρ παρακαλώ της 16. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές Απερίφθη. 22. Τμηματική σε τέσσερα μέρη. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τέταρτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Καταπίπτει. Ωραία. Ξανά. 23. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Έλεγχος. Ψηφίζουμε πρώτο τμήμα της 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, δεκτό με 16 ψήφους υπέρ. 26. Καταπίπτει. Προχωρούμε στην 25. Υπέρ παρακαλώ τις 25. Κατά. Αποχές απερίφθη. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Έλεγχος. Έλεγχος της 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 29. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 30. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 31. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 33. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Έλεγχος. Ελέγχουμε την 36, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 38 υπέρ. 37. Θα ελέγξουμε μήπως και απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε 37. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη, απερίφθη. 15 υπέρ, 15 κατά, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 40 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Έλεγχος την 40 δηλαδή, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 41. Υπέρ. Σα Κατά αποχές δεκτή. Η 42 καταπίπτει και πάμε στην 43. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος ψηφίζουμε την 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 16 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Και τώρα πάμε στην 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η έξι καταπίπτει και πάμε στην τροπολογία επτά υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Οκτώ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Έλεγχος. Η τροπολογία 8, δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Το, το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 8. Θα ξαναψηφίσουμε. Ωραία. Τροπολογία 8, δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 14 υπέρ, 15 κατά, εντάξει. Και μία αποχή. Πάμε τώρα στην τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Και Τέλος, η δέκα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και η τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Συγχαρητήρια κυρία Τόμσεν. 30 υπέρ, μία ψήφος κατά. Ε, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε κυρία Τόμψεν. Ε, ε. Επόμενο θέμα που θα ψηφίσουμε. Αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Νομίζω η κυρία Κορνέλησεν θέλει να κάνει κάποια σχόλια πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Α, κυρία η κυρία Μπραντνερ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ τώρα και η κυρία Κορνέλισεν θα την αντικαταστήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπραντνερ πριν από ένα μήνα έγινε μητέρα μιας όμορφης κόρης. Θα επανέλθει το Σεπτέμβρη και την αντικαθιστώ εγώ. Μαζί με την συνάδελφο Ουλρίκε Λούνατσεκ, όπου η Ουλρίκε είναι στην Επιτροπή Καθοδήγησης για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και διεξάγει τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό μας. Υπάρχει προσθήκη μιας πρότασης που λέει ότι οι προσλήψεις θα στηρίζεται στα αποτελέσματα και θα διασφαλίζει την ισότητα, η ισορροπία των φύλων. Καλό είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό σε Επιτροπή Γυναικών να δώσαμε σαφές μήνυμα στους εισηγητές Μπροκ και Φέρχοφστάτ ότι είναι πολύ σημαντικό για την ισότητα των φύλων και το gender mainstreaming να υπάρχουν ευθύ εξ αρχή εδρεωμένα στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Αλλιώ τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να παρεμβαίνουμε ξανά και ξανά και να λέμε ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές γυναίκες που να ε, μας εκπροσωπούν εξωτερικά, ούτε η διάσταση του φύλου λαμβάνεται υπόψη. Να ψηφίσουμε λοιπόν τις ε, τροπολογίες 4 και 5 που είναι η καρδιά της έκθεσης. Και έτσι θα δώσουμε, θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους κυρίους εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλισεν προχωρούμε στην ψηφοφορία αυτής της πολύ σημαντικής γνωμοδότησης που αφορά ε, μια εντελώς καινούρια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι πολύ σημαντικό η διάσταση του φύλου να συμπεριληφθεί ευθύς εξ αρχής. Πάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 3. Όχι, δεν θα ψηφιστεί γιατί δεν αφορά όλες τις γλώσσες, ε, τις μεταφράσεις. Πάμε στην 4. Ε, η ψήφος εδώ είναι υπέρ, Υπέρ, ε, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 7, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 8, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 9 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 1 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτό Δύο. υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας α το είπα πολύ νωρίς τώρα πέρας και εγκρίνεται 29 ψήφισαν υπέρ μια αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν και νομίζω ότι όλοι αξίζουμε συγχαρητήρια ε, για τη δουλειά μας στην ισότητα των φίλων. Συγχαρητήρια κυρία Κορνέλισεν. Ehm, Ωραία, οπότε τώρα μπορούμε να περάσουμε στην τελευταία για σήμερα ψηφοφορία. Πρόκειται την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησεις των κρατών μελών. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το Μάιο αποφασίσαμε να υποβληθούν τροπολογίες ε, στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Υπόψη της Επιτροπής Απασχόλησης. Εμείς έχουμε 35 τροπολογίες. 4 Ιουνίου έληξε η προθεσμία για την κατάθεσή τους. Επομένως ε, θα αφορά γνωμοδότηση που θα υποβάλουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, θα δώσω το λόγο σε όποιες ή όποιους συναδέλφους θέλουν το λόγο πρωτού περάσουμε στην ψηφοφορία. Κυρία Κορνέλησεν καταρχά θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι είναι κρίμα που δεν συνεδρίασαν οι Γιατί όταν εγώ κατέθεσα τροπολογίες είχα να κάνω μια πάρα πολύ ουσιαστική επιλογή. Δηλαδή, είτε να καταθέσω μια ξεχωριστή ε, γραμμή για τη διάσταση του φύλου ή να προσπαθήσω τις ε, νυν ε, γραμμές να τις τροποποιήσω. Αυτό το οποίο τελικά ε, επέλεξε ήταν να, με ένα σπάρο δύο τριγώνια, θέλετε, να σου πω να κάνω και τα δύο. Αυτό αποφάσισα. Και νομίζω ότι το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με την Επιτροπή, προς την Επιτροπή Απασχόλησης. Η κυρία Πιγκερέιδο έχει και αυτή η καταθέσει τροπολογία για μια ξεχωριστή κατευθυντήρια γραμμή. Αυτό το οποίο κάναμε είναι να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Συντάξαμε λοιπόν μια ξεχωριστή κατευθυντήρια γραμμή για τη διάσταση των φύλων και σε συνεργασία και με άλλα μέλη της Επιτροπής καταθέσαμε ξεχωριστές τροπολογίες για τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν νομίζω να υπάρξουν αντιρρήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να υπερψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες και να αποφασίσει μετά η Επιτροπή Απασχόλησης τι θέλει. Ίσως θα ήταν και μια πιο ασφαλή στρατηγική αυτή, διότι αν η Επιτροπή Απασχόληση απορρίψει την ξεχωριστή κατευθυντήρια γραμμή για τη διάσταση του φύλου, τουλάχιστον θα έχουμε τι ε, τροπολογίε που αφορούν τι εφιστάμενες κατευθυντήριε γραμμέ. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να υπερψηφιστούν όλε οι τροπολογίες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Κορνέλισεν. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω να υπάρχει κανεί Α, κυρία Μπάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση, αλλά από την άλλη πλευρά έχω και κάποιες αμφιβολίες, για να σας πω την αλήθεια. Ή ζητάμε mainstreaming, ή ζητάμε ξεχωριστό κεφάλαιο, ξεχωριστή κατευθυντήρια γραμμή, όλα ξεχωριστά. Άλλη προσέγγιση αυτή. Εγώ πάντως εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι το mainstreaming, ενσωμάτωση δηλαδή τη διάσταση του φίλου στι πολιτικέ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τι απόψεις σα. Κάποιος άλλος, αν όχι νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Περνάω στις τροπολογίες. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τροπολογία 18. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό το πρώτο. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό και το δεύτερο. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 22 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 23 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Και τώρα έχουμε μία συμβεβαστική τροπολογία, παριθμόν ένα τροπολογία συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 27 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 28 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 29 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 2 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 4 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Κύριε Φιγερέδο, ναι. Ας ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την παριθμόν 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ. Η 7 δεν απορρίφθηκε. Θέλετε να το ελέγξουμε. Ωραία, ας ελέγξουμε για το 7. It's closed and it's rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 12 αποχές. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια στην κυρία Κορνέλισεν. So, now we have to finish. Då är vi framme vid punkten 13 på föredragningslistan. Επομένως, ερχόμαστε στο σημείο 13 τα διάφορα εφόσον ολοκληρώσαμε τις ηλεκτρονικές μας ψηφοφορίες. Νομίζω ότι η συζήτηση σήμερα το πρωί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με τους εμπειρογνώμονες. Το θέμα ήταν η νεανική εγκληματικότητα και η ισότητα ανθρώπων και γυναικών υπό αυτό το πρίσμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που συνεισέφεραν στην πρωινή συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ε, τη γραμματεία. Η πρώτος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Όπως γνωρίζετε, θα ξανασυναντηθούμε άλλη μια φορά πριν ε, τις καλοκαιρινές διακοπές, ε, στα μέσα Ιουλίου, όπου θα έχουμε και την τελευταία μας συνεδρίαση. πριν το καλοκαίρι που όλοι το περιμένουμε τόσο πολύ. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν στη συνεδρίαση της Επιτροπής τον Ιούλιο. Ευχαριστώ πολύ.